Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έχουμε στην μέση διάταξη σήμερα την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας καλωσορίζω σε αυτή την ευχάριστη αίθουσα συνεδριάσεων. Πριν δώσω το λόγο στον συγκητή, θα καλωσορίσω την Επίτροπο ε, Κούγεν Κουίν ε, αρμόδια για θέματα έρευνας και πάλι καλώς ορίσατε ε, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Το γεγονός ότι σας ξανακαλέσαμε δείχνει ότι είναι πολύ σημαντική για μας η έρευνα και στον προπολογισμό της Ένωσης και σας ευχαριστώ που ήρθατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις της Επιτροπής μας. τα διαδικαστικά πρώτα. Έγκριση μερίσια διάταξη. Δεν βλέπω κανένα να επιθυμεί αλλαγή τη, οπότε θεωρώ ότι το σχέδιο εγκρίνεται όπω σα έχει διανεμηθεί. Επιπλέον να σα πω ότι είναι δημόσια η συνεδρίαση και μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Και ότι η ε, μετάφραση επίσης είναι στη διάθεσή σας. Και ευχαριστώ και τις μεταφραστικές υπηρεσίες. Λοιπόν... Έρχομαι στο σημείο 3 αμέσω τη σημερινή ημέρα διάταξη και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μάρκους Πίπερ για τις εισαγωγικέ παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε καθυστέρηση 13 λεπτά. Ίσως θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη ε, πειθαρχία στις συνεδριάσεις εφόσον θέλουμε να έχουμε και ακρίβεια στη διαδικασία απαλλαγή. Κυρία Επίτροπε, Καλώ ήλθατε κυρία Γκέγον. Γκίγαν Κουίν, κύριε Μπάλκο από το Ελεκτικό Συνέδριο, αγαπητοί συνάδελφοι, το ποσοστό των σφαλμάτων που έχουμε στον τομέα της έρευνας και στα συναφή θέματα βρίσκεται το 2012 στο 3,9% και λόγω των νέων μεθόδων ε, υπολογισμού του ελεγκτικού συνεδρίου που αλλάζει την, τον υπολογισμό φτάνουμε σε 2,1% ποσοστό ε, σφαλμάτων. Βρισκόμαστε λοιπόν στο κατόφλι της σημαντικότητος σε ό,τι αφορά τα σφάλματα και γι' αυτό θέλω να εκφράσω την ε, αναγνώρισή μου για το γεγονός αυτό. Το ελεκτικό συνέδριο στην έκθεσή του υπογραμμίζει την, την υψηλή ποιότητα της δράσης της Γενικής Διεθνής Έρευνας και Καινοτομίας. Πράγματι, είναι πολύ καλή η παρουσίαση των στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης. Δεν χρησιμοποιεί κορακίστικα όπως σε άλλες γενικές διευθύνσεις. Ο τομέας της ε, έρευνας υπόκειται σε συγκεντρωτική διαχείριση, είναι η Κομισιόν αρμόδια για την ε, διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά τα κονδύλια. Αλλά, εδώ πρέπει να σταθώ πιο επικριτικός, εδώ και πολλά χρόνια εξακολουθούν να υπάρχουν σφάλματα, υπάρχουν κονδύλια τα οποία δεν θα έπρεπε να λαμβάνονται από τους ε, δικαιούχους και εδώ και δεκαετίες λέει η Κομισιόν ότι θα βελτιώσει την ε, ε, πληροφόρηση προς τους δικαιούχους και με σεμινάρια θα τους εκπαιδεύσει καλύτερα για τις ανάγκες σαφήνεια στα κονδύλια αυτά και το τι καλύπτουν. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες από την Κομισιόν και θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν έχετε κατά κάποιο τρόπο ένα κατάλογο κατά σφαλματούχων, αν υπάρχουν ε, σε ορισμένα σχέδια περισσότερα σφάλματα, υπάρχουν χώρες όπου είναι περισσότερα τα σφάλματα από άλλα και αυτά που θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε κάποια σκέψη. Μήπως λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε αν θα πρέπει να μην περιλαμβάνονται ορισμένοι χώροι λόγω του υψηλού, στη χρηματοδότηση λόγω του υψηλού ποσοστού φαρμάτων. Η Κομισιόν έχει απλοποιήσει βέβαια μετά από κατά αποκόπη την διαχείριση αλλά και τους ελέγχους εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Το ερώτημα είναι όμως αν θα μπορούσαμε να έχουμε και μία ενημερωμένη έκθεση της Κομισιόν που να περιλαμβάνει και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή τις ε, απλοποιημένες διαδικασίες ήδη για το 2012. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε και αυτά τα στοιχεία εν ώψη της ε, Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν τις επόμενες μέρες μπορούμε ήδη να έχουμε αυτές τις ανακοινώσεις από την Κομισιόν για το θέμα αυτό, για το κατά πόσο ήταν επιτυχής η διαδικασία αυτή απλοποίησης. Αν λοιπόν η Κομισιόν με τον τρόπο αυτό είδε να υπάρχει αύξηση, μάλλον υπολογίζω θα υπάρξει αύξηση του ποσοστού σφαλμάτων ή όχι. Και εάν υπάρξει αύξηση των σφαλμάτων λόγω της απορροπήσης, πού θα βρίσκεται το πρόβλημα που θα οδηγήσει τα σφάλματα. Δύο ακόμα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλές γενικές διευθύνσεις οι οποίες εμπλέκονται στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Οπότε υπάρχει κάποια δυσκολία διαχείρισης λόγω αυτού Ίσως, κύριε Πίτροπε, θα μπορούσατε εν συντομία να μας εξηγήσετε πώς βλέπετε το θέμα του συντονισμού μεταξύ των γενικών διευθύνσεων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα έρευνας, ώστε να μην υπάρξει αυτό αιτία τριβών και προβλημάτων. Το τελευταίο ερώτημά μου προς την ε, κυρία Πίτροπο αφορά το το ΙΤΕΡ και την κατανομή αρμοδιοτήτων σε σχέση αυτό. Πώς γίνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιτρόπων και υπηρεσιών. Αυτά είναι τα ερωτήματά μας που είναι περιορισμένα βέβαια. Έχουμε υποβάλει πολλά ερωτήματα στην ε, κυρία Επίτροπο και περιμένουμε να ακούσουμε και τη θέση της κυρίας Επιτρόπου αλλά φυσικά και τη θέση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή με την συντομία σας ε, μας έχετε εξοικονομήσει και χρόνο ώστε μειώνεται η καθυστέρηση η οποία οφείλεται στα μεταφορικά μέσα και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Σλαβ Μπάλκο από το Ελεκτικό Συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ κύριε τώρα. Αγαπητή Πρόεδρε τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, κύριε Σιγητά, κύριε Πίπερ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Αγγίγκαν Κουίν, Κυρίες και κύριοι. Uh, Πριν από δυόμισι μήνες και κάτι, σας παρουσίασα την ειδική έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου ε, υπαριθμών 2 του 2013 για τον... Ε, έλεγχο της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής ε, του ε, προϋπολογισμού και σήμερα θα σας πω κυρίως ε, τα της εφαρμογής του 7ου προγράμματος πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα το κεφάλαιο 8 της ετήσιας έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου για το 2012 που αναφέρεται κυρίως στη διαχείριση των δαπανών για την έρευνα. Τα ερευνητικά προγράμματα αποτελούν την προτεραιότητα των δαπανών που ε, άπτονται αυτού του κεφαλαίου και πιο συγκεκριμένα το 68%. Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, ο βασικός κίνδυλος παρατυπιών είναι το γεγονός ότι οι δικαιούχοι μπορεί να συμπεριλάβουν ε, μη επιλάξιες δαπάνες ή δαπάνες οι οποίες δεν αιτιολογούνται δεόντως και αυτά ε, δεν διορθώνονται από τα υποπτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κίνδυνος αυτός ε, διωγγώνεται από τον ε, κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τον τρόπο υπολογισμού του κόστους, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει και τώρα. Γι' αυτό λοιπόν τα μέτρα τα οποία εισάγονται από την απόφαση της Επιτροπής του Ιανουαρίου του 2011 για την απλούστευση των κανόνων για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο θεωρούμε ότι συνεισέφεραν στη μίεση του διοικητικού άχθους για τους δικαιούχους και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον έλεγχο που έγινε ε, για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο από τις μεθοδολογίες που χρησιμοποίησαν για τον έλεγχο. and Αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα και θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω απλούστευση ε, η οποία θα προέλθει μόνο από τον ορίζοντα 2020, κάτι το οποίο ε, εγκρίνατε εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από δύο εβδομάδες και την Τρίτη εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο. Το ελεγκτικό συνέδριο στη γνωμοδότηση 6 του 2012 υποστήριξε την έγκριση αυτών των κανόνων για τον ορίζοντα 2020, για τη συμμετοχή στα νέα ερευνητικά προγράμματα για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ποια είναι τα βασικά λοιπόν μηνύματα τα οποία αφορούν ε, τις ε, ερευνητικές δαπάνες για το 2012. Καταρχάς, Όσον αφορά ε, το αν είναι ε, νομότυπες ε, οι συναλλαγές στο σύνολό τους, ο έλεγχος, ο δειγματοληπτικός που έκανε το ελεγκτικό συνέδριο, διαπίστωσε ότι 49% περιλαμβάνουν σφάλματα και όπως είπε και ο κύριος Πίπερ, το ποσοστό σφάλματα είναι της τάξης του 3,9% που είναι υψηλότερο από το 3% που είχαμε το 2011, αλλά αυτό θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε ε, και από την αλλαγή του τρόπου που λαμβάνει δείγματα το ελεγκτικό συνέδριο, όπως εξήγησε και η κυρία Κελουλάρ και ο συνάδελφος David Μπός την προηγούμενη εβδομάδα, όταν παρουσίασαν το κεφάλαιο 7 για την ε, βοήθεια της εξωτερικές σχέσεις και την ε, διεύρυνση. Στο κεφάλαιο 8, οι πιθανότητες φάλματος δείχνουν ένα 62% και θεωρούμε ότι έχουμε συνεισφορά μίας ποσοστίας μονάδας, όπως αναφέρθηκε και από τον εισηγητή. Το βασικότερο πεδίο σφαλμάτων είναι το γεγονός ότι έχουμε μη επιλέξιμες δαπάνες και επειδή χρησιμοποιούνται ε, λανθασμένες μέθοδοι υπολογισμού από τους δικαιούχους για τα προσωπικά και για τα έμεσα κόστη και πάλι έχουμε σφάλματα. Το ελεγκτικό συνεργείο διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις το 2012 όπου οι συντονιστές των προγραμμάτων ε, ε, ενθάρρυναν τις μακροχρόνιες καθυστερήσεις ε, και επειδή αυτές οι καθυστερήσεις μπορεί να έχουν πολύ σημαντικές οικονομικές συνέπειες, κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ελεγκτικό συνέδριο κάνει μια νέα σύσταση πολύ συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τέταρτον, το συνέδριο θεώρησε ότι τα νέα συστήματα ελέγχου είναι εν μέρει αποτελεσματικά και θεωρούνται εν μέρει αποτελεσματικά διότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες στους ελέγχους δεν διαπιστώθηκαν σφάλματα ε, στις πληροφορίες που υποβάλλουν οι δικαιούχοι. Τα πιστοποιητικά βέβαια τα οποία δίνονται από ανεξάρτητους ελεγκτές ε, και αυτά θεωρήθηκαν ότι είναι εν μέρει αποτελεσματικά. Παρά το γεγονός ότι το συνέδριο αναγνωρίζει ότι ε, αυτές οι μέθοδοι βοηθούν ίσως να μειώσουν τον αριθμό των σφαλμάτων για το 7 πρόγραμμα πλαίσιο, ε, διαπιστώνουν πολλές φορές ότι υπάρχουν αρκετά σφάλματα στις δηλώσεις για τις δαπάνες οι οποίες είναι πιστοποιημένες από ανεξάρτητους ελεγκτές. Αυτό το είδαμε στις 29 από τις 35 δηλώσεις που υπευλήθησαν. Η έλεγχη είναι αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος ελέγχου, αλλά όπως υπάρχει το νέο σύστημα, ε, δεν μας βοηθά να μειώσουμε τα σφάλματα. Είναι σχεδιασμένο για να μας δίνει διασφαλίσεις σε πολιετές πλαίσιο μειώνοντας ε, το ποσοστά ασφάλματος ε, για τα ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, το ελεγκτικό συνέδριο αναθεώρησε και τους ε, στρατηγικές ελέγχου των διαφόρων γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής και διαπίστωσε ότι το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Όργανο και οι άλλοι ελεγκτικοί οργανισμοί δεν θεωρούν ότι εφαρμόζουν ικανοποιητικά τους ελέγχους και για το 7ο και για το 6ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο διαπίστωσαν 1.700 περιπτώσεις ε, σφαλμάτων ε, που θεώρησαν ότι υπάρχουν σφάλματα τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν και πάνω από 1.400 περιπτώσεις πρέπει ακόμα να διορθωθούν βάσει των πληροφοριών που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα έχουμε πάνω από 800 ακόμα περιπτώσεις που βασίζονται σε ελέγχους που έγιναν το 2011. Και το ελεγκτικό συνέδριο κάνει και σχετική σύσταση. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων ε, διαφόρων ε, ανεξαρτήτων οργανισμών και αποκεντρωμένων οργανισμών μας δίνουν αρκετά στοιχεία για ε, τις παρατυπίες που έχουμε στις ετήσιες συναλλαγές. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων ε, του Οργανισμού Έρευνας και Ανάπτυξης αποτελεί ένα καλό παράδειγμα καλής πρακτικής. Οι συστάσει ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ελεκτικού Συνεδρίου είναι αντίστοιχε με αυτέ που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε επίσης μια επιπλέον σύσταση να μην σταματήσουν τις προσπάθειές τους για να μπορέσουν να μειώσουν τα σφάλματα τα οποία διαπιστώνονται και επίσης να υπενθυμίσουν στους δικαιούχους και στους ελεκτέ ποιοι είναι οι κατάλληλοι κανόνες για τις επιλέξιμες δαπάνες. Και επίσης θα πρέπει οι συντονιστές των προγραμμάτων ε, να ε, διανέμουν τις δαπάνε, τα κονδύλια το συντομότερο δυνατόν και εάν γίνεται, υπάρχει ανάγκη για οποιαδήποτε τροποποίηση να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις καθυστερήσεις, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ούτε για τον, τους ε, εκτονιστέρων των ελέγχων, ούτε για τις περιπτώσεις στις οποίες γίνεται παρεκβολή των αποτελεσμάτων. Όλες αυτές οι στάσεις θεωρούνται θετικές να ευχαριστήσω την κυρία Γκέγκαν Κουίν και τους συναδέλφους της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικοδομητική συνεργασία και με εμά και με εσά. Και να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προσοχή του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπάλκο. Είστε μέλο του ελεγκτικού συνεδρίου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, εξηγήσει αυτέ και την παρουσίαση, την ετήσια έκθεση και θα παρακαλέσω την αξιότιμη κυρία Επίτροπο να μα παρουσιάσει ε, τη δική της ε, άποψη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Πίπερ, ε, αντιπρόεδροι, αξιότιμα μέλη, κύριε Πάλκο, συνάδελφοι. Με χαρά έχουμε ξανά στην Επιτροπή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2012. Έχουμε την ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, και τώρα ε, πρέπει να συζητήσουμε για την ερευνητική πολιτική. Κάποια εισαγωγικά σχόλια. Χαίρομαι που το Συμβούλιο Υπουργών αυτή την εβδομάδα ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενέκρινε επίσημα το νομοθετικό πακέτο για τον ορίζοντα 2020. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι εκ των όνου κάνευ προαπαιτούμενα ε, για την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση τη οικονομία, την καταπολέμηση τη ανεργία και γενικότερα τι προκλήσει που έχουμε στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι το πρόγραμμα Ορίζον 2020 ε, δίνει την έμφαση σε προγράμματα και σχέδια για συγκεκριμένα ερευνητικά αποτελέσματα για την καινοτομία ε, με οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Και εσείς ο ίδιος κύριε Πρόεδρε κάνετε μια αντίστοιχη έκθεση αξιολογώντας τα οικονομικά ε, ε, της Ένωσης σε σχέση με τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει. Δεν θα πρέπει να υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατική επιβάρυνση. Έρχομαι στο δεύτερο χαρακτηριστικό ε, του ορίζοντα 2020 που είναι πολύ προσφυλής και στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή σας και σε μένα. Η απλούστευση για τους δικαιούχους. Είναι ε, γενικά ε, αυτά τα θέματα και επιταγές να μπω σε πιο ε, επιμέρους θέματα. 3,9% ακούσαμε για τα σφάλματα, υψηλότερο ποσοστό από ό,τι πέρσι, αλλά όπως λέγει και το ίδιο το συνέδριο αλλά και ο εισηγητής, στην παράγραφο 813 της ετήσιας έκθεσης, αυτό οφείλεται κυρίως στην αλλαγή της μεθοδολογίας που ακολουθεί το ελεκτικό συνέδριο. Σε ό,τι αφορά την έρευνα, το ελεκτικό συνέδριο δίνει μια εικόνα για το σύνομο και τις παρατυπίες ε, και αυτό... Ε, ε, έρχεται να επικυρωθεί και από τα δικά μας ευρήματα που το εκτιμούμε γύρω στο 5% ε, μειώθηκε ε, σε 3,5 με 4% μετά από τις διορθώσεις και τις ανακτήσεις να έχουν ληφθεί υπόψη. Η πηγή του σφάλματος παραμένει σε όλες τις κατηγορίες και σε όλους τους δικαιούχους παρόλο που δείχνουν ότι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι δικαιούχοι κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν σε σφάλματα. Οπότε ερώτημα. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περιορίζει τον αριθμό σφαλμάτων που παρατηρούνται. Πρώτον, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της ε, περίοδου του 7ου προγράμματος πλαισίου, προχωρούμε ε, σε λύσεις, όχι όμως βραχυπρόθεσμες, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τώρα στο τέλος του προγράμματος για τόσο λίγο χρόνο. Βελτιώνουμε όμως τις ε, διαδικασίες συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων εκ των προτέρων για να μειώνονται τα σφάλματα, να μειώνεται και ο χρόνος που χρειάζεται από την αρχή, από την ε, διαπραγμάτευση ε, την υπογραφή των συμβάσεων μέχρι την πληρωμή των δικαιούχων. Αυτό είναι μια διαρκής διαδικασία. Προσπαθούμε να είναι πιο προσαρμοσμένα στις ανάγκες των δικαιούχων τα προγράμματα, ανεξάρτητοι οι ελεγκτές ε, ε, και το προσωπικό μας από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας έχουν κάνει συνολικά 24 παρουσιάσεις σε χώρες μέλη και συνδεδεμένες φέτος μόνο και με 3.100 ε, ε, παραλήπτες αυτής της ε, ενημερωτικής εκστρατείας που είχε πάρα πολύ καλή απήχηση και αυτό απαντά και στις ανησυχίες του ελεκτικού συνεδρίου ως προς την ποιότητα των πιστοποιητικών ελέγχων. Επίσης συνεχίζουμε να κάνουμε ελέγχους εκ των υστέρων και ανακτήσεις όπου έχουμε το καταβληθέντα ποστά και αυτό το έχουν διαπιστώσει είτε οι δικοί μας υπάλληλοι είτε του ελεκτικού συνεδρίου. Έτσι θα μειωθεί το υπόλοιπο, οπότε δεν χρειάζεται επιπλέον ε, οι ερευνητές να επιβαρύνονται με διοικητικό άκθος, δηλαδή να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των ελέγχων ή να ζητούμε όλο και περισσότερες πληροφορίες πριν την καταβολή των πληρωμών. Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι προσιλωμένη στην προσπάθεια αυτή, συνεχώς θα αναθεωρούμε και θα βελτιώνουμε τα ε, συστήματά μας για να παραμείνει όσο γίνεται χαμηλότερος ο αριθμός σφαλμάτων. Για το μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να μειωθεί το ποσοστό σφαλμάτων ιδιαίτερα με απλουστεύσεις στο ορίζον 2020. Για το έμεσο κόστος ένα καλό παράδειγμα είναι ένα καταποκοπή ε, ποσό οι ε, δικοί μας ελεκτές αλλά και του ελεκτικού συνεδρίου βλέπουν ότι υπάρχουν σφάλματα στη δήλωση του εμέσου κόστος. Αυτό θα σταματήσει στον ορίζοντα 2020 και άλλες απλουστεύσεις έχουν να κάνουν με ένα ενιαίο συντελεστή βοήθεια για όλους τους ε, δικαιούχους με σαφείς κανόνες για το, ε, τις διοικητικές δαπάνες με περισσότερη ελαστικοποίηση, εξωτερική ανάθεση, υπεργολαβίες κτλ. Αυτό στην γνωμοδότηση 6 του 2012 αναφέρεται για τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης ε, στο πρόγραμμα Horizon 2020. Αποφεύγουμε μια μεγάλη πηγή σφαλμάτων που είναι το έμεσο κόστος βέβαια παραμένει κάποιος κίνδυνος και αναπόφευκτος είναι αυτός ουσιαστικά βασικός και γενικός κανόνας για πληρωμές θα ε, είναι βάση παραστατικών και πραγματικών δαπανών ε, αποζημίωση ε, και θα απαντά στις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων. Με μια τέτοια χρηματοδότηση υπάρχει αναπόφευκτος κίνδυνος φαλμάτων και το έχει επισημάνει αυτό το ελεκτικό συνέδριο. Δεύτερον, στην ετήσια έκθεσή του για το 2012 ο Γενικό Διευθυντή Έρευνα και κοινοτομία δήλωσε ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει έχουν διπλάσιο του μέσου όρου σφάλμα και τριπλάσιο είναι εκείνο των νέων δικαιούχων που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Κανεί δεν θέλει όμω να αποκλείσει τι μικρομεσαίε ή του νέου δικαιούχου εκτό του προγράμματο, μόνο και μόνο για να ελέγχουμε το ποσοστό σφαλμάτων. Συμφωνούμε και τα τρία θεσμικά όργανα ότι χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη στι μικρομεσαίε και είναι ουσιαστικότατη για να αυξηθεί η καινοτομία στην Ένωση και θα πρέπει να ανοίγουν τα προγράμματα σε νέου συμμετέχοντε για να καλύπτεται το ερευνητικό πεδίο παντού στην Ευρώπη. Ε, αυτό συνοδεύεται και από ένα υψηλό κίνδυνο σφάλματο, αλλά αξίζει τον κόπο να το ε, ρίψω κινδυνεύσουμε. Ε, είναι πολύ σχεδής αυτή η διαδικασία και ε, περίπλοκη, αλλά είναι απαραίτητη για να δημιουργούνται θέσει εργασία στην Ευρώπη και κάποιο κίνδυνο θα πρέπει να παίρνουμε, εάν θέλουμε σοβαρά να φτάσουμε σε αυτού του στόχου. Είναι πρόκληση να παραμείνει σε ένα αποδεκτό επίπεδο το σφάλμα χωρίς αυτό να είναι εις βάρος μιας ουσιαστικής ε, ερευνητικής πολιτικής. Είμαι πεπισμένη ότι ο ορίζον 2020 θα είναι καμπή πραγματική για να έχουμε ε, απλές επενδύσεις δίκαιες και σωστές πανευρωπαϊκά στην έρευνα. Οι προτάσεις επίσης θα μας ε, βοηθήσουν να φροντίζουμε κάθε ευρώ να πιάνει τόπο γιατί το ζητούν οι φορολογούμενοι και το αξίζουν ε, οι επενδύσεις τους να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Συμπερασματικά σας διατρανώνω και πάλι την προσήλωσή μου στην υγιή ε, διαχείριση των οικονομικών. Υποστηρίζουμε την αριστεία στην έρευνα, την καινοτομία ε, με επενδύσεις και πολιτική ελκυστική για να επενδύουμε σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη της οικονομίας αισιόδοξη ότι θα βρούμε τη σωστή ισορροπία, τη χρυσή τομή και θα φτάσουμε και στους δύο στόχους στο επόμενο διάστημα, στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και στη συνέχεια με τον ορίζοντα 2020. Ξέρω ότι ο κύριος Πίπερ έκανε μια σειρά συγκεκριμένων ερωτήσεων στις οποίες θα απαντήσω, αλλά νόμιζα καλύτερα ήταν να κάνω την εισαγωγή μου και στη συνέχεια να απαντήσω και στις υπόλοιπες ερωτήσεις που θα κάνουν και άλλα μέλη της Επιτροπής. Εάν το δέχεστε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κιγκον Κουίν για τη δήλωσή σας και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη στην προσέγγιση επί τη βάση σχολείων για την, ε, μέσω της εκθέσης ε, στην οποία εγώ είμαι εισηγητής θα προσβλέπω στη συνεργασία μας αγαπητοί συνάδελφοι τώρα περνάμε στην, στον διάλογο με την ε, κυρία Επίτροπο Υπάρχουν τώρα συνάδελφοι οι οποίοι θα θέλαν να λάβουν το λόγο. Η κυρία Προζομπάτα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με τις ε, ενέργειες που είχαν υψηλό επίπεδο κινδύνων. Τι είδους ε, ε, τέτοιες ε, διαδικασίες είχαν, επέχουν υψηλό επίπεδο κινδύνου. Ο Γιάν Μίλντερ ακολουθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως μπορεί να είναι παρηγοριά για μας για, για τους υπευθύνους της Κομισιόν στον τομέα αυτό ότι το ποσοστό σφαλμάτων είναι, είναι χαμηλότερο από το μέσον όρο των σφαλμάτων σε όλο τον προπολογισμό και αυτό εν του γεγονότος τα προγράμματα αυτά είναι πολύ πεπλεγμένα και είναι πάρα πολλά τα μεμονωμένα συμβόλαια και οι συμβάσεις. Το ερώτημα μου στρέφεται προς το ελεκτικό συνέδριο και προς την Επίτροπο. Έχουν γίνει διορθώσεις σε οικονομικό επίπεδο. Εάν μιλάμε για το ποσοστό σφαλμάτων, εκεί περιλαμβάνονται και οι διορθώσεις ή όχι. Και αν περιλαμβάνονται οι διορθώσεις γιατί δεν αναφέρεται αυτό όπως έχει τώρα η έκθεση. Το δεύτερο ερώτημα είναι είναι ρεαλιστικό να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα μέσον όρο 2%. Κάθε χρόνο βλέπουμε γιατί δεν επετεύχθη αυτό το 2% και συζητάμε τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση αλλά αυτή είναι η 19η φορά που δεν έχουμε φτάσει το 2% μόνο. Υπάρχει η πιθανότητα να φτάσουμε αυτό το στόχο ή πρέπει να πει η Κομισιόν ότι ο στόχος του 2% είναι μη ρεαλιστικός και πρέπει να θέσουμε ένα διαφορετικό στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω καταρχήν την, ε, το Ελεκτικό Συνέδριο και την κυρία Επίτροπο για τις παρουσιάσεις τους. <clears throat> Μας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Προσπαθούμε να στρέψουμε τα μάτια μας προς το μέλλον και θέλουμε να δούμε πώς θα αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρήσεών τους. Θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου το εξής. Ο τομέας αυτός της έκθεσης 2012 για την απαλλαγή περιλαμβάνει μια συχνότητα σφαλμάτων 49% όπως και στην κοινή αγροτική πολιτική. Θα ήθελα να ξέρω αν αυτή η νέα μεθοδολογία έχει επηρεάσει το ποσοστό σφαλμάτων που είναι 30%. Μας είπε τώρα το ελεκτικό συνέδριο ότι έχει αλλάξει μεθοδολογία και πρέπει να προσθέσουμε και κάτι σε σχέση με τις υποκαταβολές το οποίο δεν εμφανίζεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το 49% το οποίο αναφέρθηκε επίσης ως ποσοστό οφείλεται και αυτό στη νέα μεθοδολογία. Θα ήθελα να πω ότι κατανοώ αυτά τα οποία ελέγχθηκαν, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το ελεκτικό συνέδριο αν είναι αξιόπιστη αυτή η αριθμή, αν υπάρχει πρόβλημα μεθοδολογίας. Προς την Επίτροπο, ο Ισπανικός τύπος έχει γράψει ότι υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των δικαιούχων αν θα, θα, μετά από αυτά που δημοσιεύτηκε, δηλαδή, θα ήθελα να υπάρχει ένας κατάλογος των δικαιούχων στους διάφορους τομείς δράσης σας. Έχουμε ενέργειες βέβαια που περιλαμβάνουν κόστος το οποίο δεν μπορεί να υπολογιστεί σωστά και μεθοδολογία που δεν εφαρμόζεται. Αλλά αν δούμε το τομέα της καινοτομίας, ποιοι είναι οι τομείς που δείχνουν να έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο και πού μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση εν του ορίζοντα 2020. Επίσης, αναφέρεται και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο νότιο μέρος της Ευρώπης αλλά και στο βόρειο λιγάκι. Το πρόβλημα της πληρωμής προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει βελτιωθεί λοιπόν το θέμα αυτό, η καθυστερήσει προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα μπορέσουμε με τον ορίζοντα 2020 να βάλουμε πάγο στις καθυστερήσεις αυτές που παρουσιάζονται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προσπαθούμε βέβαια με όλα τα μέτρα να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά υπάρχουν και διαμαρτυρίες από τους δικαιούχους που λένε ότι δεν υπάρχει ευκαμψία, επαρκής ευκαμψίας σε ένα τόσο πολυδέδαλο και πολύπλοκο τομέα και είναι δύσκολο για αυτούς να αλλάξουν ε, να προσαρμοστούν σε αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει στην, ε, στην ε, αρχική σχεδίαση. Θα ήθελα να ξέρω αν έχει βελτιωθεί λοιπόν αυτή η κατάσταση με τις αλλαγές που επέφερε η Κομισιόν. Και παρόλα αυτά θέλω να συγχαρώ την Επίτροπο γιατί υπήρξαν σίγουρα βελτιώσεις στα συστήματα και στην ετήσια έκθεση είναι η καλύτερη εκθέση που έχουμε δει μέχρι στιγμής και μπορεί να θεωρηθεί βέλτιστη πρακτική. Ευχαριστώ πολύ. Η Ανδρέασεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα αναφερθώ σε αυτή τη συχνότητα 49% σφαλμάτων στον αριθμό των συναλλαγών που ελέγχθησαν από το ελεγκτικό συνεδρίο. Εάν παίρνουμε ένα δείγμα και το 50% των συναλλαγών έχει πρόβλημα, αυτό δημιουργεί πολύ κακή εντύπωση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται κανείς το πρόγραμμα. Μήπως θα μπορούσε να μας εξηγήσει Επίτροπος πώς θα αντιμετωπίσει το ορίζον 2020 αυτό το πρόβλημα. Πώς σκοπεύει να περιορίσει τη συχνότητα σφαλμάτων στις συναλλαγές. Διότι ε, το να μιλάμε απλώς για την απλούστευση των κανόνων είναι κάτι το οποίο το κάνουμε εδώ και 10 χρόνια. Και έχω την εντύπωση ότι όλες οι απλουστεύσεις που έχουν εφαρμοστεί δεν αρκούν. Θέλω λοιπόν μια πολύ απλή εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο το Horizon 2020 θα επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Και με βάση αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε και το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από ό,τι φαίνεται, το σφάλμα το οποίο παρουσιάζουν κατά μέσο όρο είναι το διπλάσιο των υπόλοιπων πολιτικών. Και πού έγκυται αυτό το ποσοστό σφάλματος. Το σφάλμα είναι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κανονισμό της. Και εδώ ερχόμαστε πάλι στον τρόπο με τον οποίο απαντάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι απλώς θα πλουστεύσουμε τους κανόνες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται συγκεκριμένη προσοχή εδώ, διότι αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μέτρα λοιπόν μπορούν να ληφθούν συγκεκριμένα για αυτές τις επιχειρήσεις. Ja, vielen Dank, äh, Frau Andreasen. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Ανδρέασεν. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση που συνδέεται με αυτό που μόλις είπε η κυρία Ανδρέασεν. Κύριε Επίτροπε, εσείς ε, ε αναφέρετε ότι οι απροστεύσεις που κάνατε στον ορίζοντα 2020, κατά την άποψή σας, θα οδηγήσουν σε μείωση ε, του αριθμού των σφαλμάτων ή του ποσοστού. Όταν το συζητάει κανείς με μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, ε, πάντα μας επιπλήττουν ότι είναι δύσκολες οι διαδικασίες λένε και πρόσφατα σε μία εκδήλωση μας είπαν ότι δεν υπάρχουν ε, ε, οι κανόνες σε όλες τις γλώσσες και επίσης διαμαρτύρονται και καταγγέλουν ότι ορισμένοι κανόνες αλλάζουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ερώτηση. Πώς απαντάτε σε αυτές τις αιτιάσεις, μπορείτε είναι υπόψη σας, τις γνωρίζετε και ποια βήματα επιθυμείτε να κάνετε έτσι ώστε στο μέλλον έτσι να υπάρχει και μια αξιόπιστη ρύθμιση και κανόνες που να ισχύουν για την περίοδο ας πούμε 2014-2020 θα εκδώσετε κανένα εγχειρίδιο ηλεκτρονικά δεν λέω να μπορεί κανείς να κατεβάζει αν θέλει να υποβάλει μια αίτηση και ε, με δεσμευτικούς ορισμούς ε, των ε, διαφόρων νομικών ορισμών και ενιών για να μπορούν να απευθύνονται εκεί αξιόπιστα οι ενδιαφερόμενοι. Ο κύριος Πίπερ, ο εισηγητής, έχει ερωτήσεις. Οι συνάδελφοι με κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό και τα κενιά που υπήρχαν. Υπήρχε κάτι που ήταν ένα σειρμός σε όλη αυτή τη συζήτηση που είναι η σύγκρουση μεταξύ Ελεκτικού Συνεδρίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις ε, flat rates, έτσι, τις καταποκοπή διορθώσεις που τελικά μπορεί να επηρεάσουν το ποσοστό των σπαλαμάτων αλλά μπορεί και όχι. Εγώ δεν θέλω να μεροληπτήσω ή να πάρω θέση, αλλά θα ήθελα να μου πούν πώς το αξιολογούν Ελεκτικό Συνέδριο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μήπως υπάρχει έδαφος εκεί να ε, προσεγγιστούν οι απόψεις. Άλλος δεν θέλει... Α, η κυρία Γιάλα κάτι ξέχασε. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Σε σχέση με αυτό που έλεγε ο εισηγητής, ο κύριος Πίπερ, για τις κατακοπήν διορθώσεις, θα ήθελα κι εγώ να ξέρω μέχρι ποιο βαθμού μπορεί ο εκ των υστέρων μηχανισμός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να εντοπίσει κάποια από τα προβλήματα τα οποία ε, υπάρχουν τόσο για τους εκ των υστέρων και όσο για τους εκ των προτέρων ελέγχων, τουλάχιστον με βάση τα όσα μας λέει ο εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου. Κατά πόσο λοιπόν αυτές ε, οι αποκοπήν διορθώσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέσο απλούστευσης και να αλλάξει και ο τρόπος που τα αντιλαμβάνονται όλα αυτά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μειώσουμε και το κίνδυνο σφάλματος στο μέλλον. Εγώ συμφωνώ καταρχήν αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σε περίπτωση λοιπόν που διαπιστωθούν εκ των υστέρων προβλήματα σε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε αυτά να τα διορθώσουμε βραχυπρόθεσμα. Τι μπορούμε να έχουμε στον νέο ορίζοντα 2020 γι' αυτό. Ja, vielen Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Επίτροπο να απαντήσει στο βαθμό του δυνατού τα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολλέ οι ερωτήσει οι οποίε διατυπώθηκαν, αλλά υπάρχει και ένας μύτος ο οποίος διατρέχει όλες αυτές τις ερωτήσεις που θα με βοηθήσει να απαντήσω. Αν μπορώ να σας απαντήσω χωρίς να ακολουθώ τη σειρά που τέθηκαν. Γιατί δεν έχουμε ένα εγχειρίδιο που να δίδεται στους εμπλεκομένους. Θα έχουμε ένα εγχειρίδιο για δημοσιονομικές ε, διαδικασίες στην δικτυακή πύλη του ορίζοντα 2020. Με την εμπειρία που έχουμε θα είναι πιο φιλικό προς τους χρήστες. Θα μπορούν να καταλαβαίνουν καλύτερα οι εμπλεκόμενοι στα προγράμματα τι πρέπει να κάνουν από ό,τι στο παρελθόν, αλλά αυτό το εγχειρίδιο, το εγκόλπιο αυτό, θα έχει το χαρακτήρα το καταλόγου των δημοσιονομικών ε, κανόνων. Ε, ο εισηγητής θέλει να ξέρει τι κάνουμε με αυτούς οι οποίοι κατ' επανάληψη έχουν κάνει ε, ατασταλίες ή σφάλματα. Όταν έχουμε να κάνουμε με διαδικασίες ανάκτησης, ιδίως σε μεγάλους οργανισμούς, νομίζω όλα αυτά τα οποία γίνονται ε, έχουν αποτέλεσμα στο μέλλον και μας επιτρέπουν να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε περιοχές που υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Υπάρχουν και τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλουμε, τα οποία θα φτάσουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ το 2012. Επίσης, πολλοί βουλευτές έθεσαν το ερώτημα γιατί υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες στο ε, πρόγραμμα πλαίσιο 7 ή αν διαφορετικής ερμηνείας και τι κάνουν στον ορίζοντα 2020 που θα εμποδίσει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αυτό το ερώτημα πράγματι τέθηκε πέρσι όταν ήμουν εδώ μαζί σας για την απαλλαγή. Στον, ε, στον ορίζοντα 2020 θα έχουμε ένα κοινό κέντρο υποστήριξης το οποίο θα καλύπτεται από τη Γενική Διεθνής Έρευνα και Κοινοτομίας, θα είναι κοινό και για επιχειρηματικέ δραστηριότητε, για έλεγχο, για νομικά θέματα και για πληροφορική. Με τον τρόπο αυτό θα φτιάξουμε μια καλύτερη απάντηση και θα μπορούμε να έχουμε και μια πιο συνεκτική εικόνα όλων αυτών που λαμβάνουν χώρα και δεν θα είμαστε στην ίδια κατάσταση που είμαστε στο παρελθόν όπου αν εξαρτιόταν από ποια γενική διεύθυνση εξαρτιέστε ή από ποιον υπάλληλο της γενικής διεύθυνσης που μπορούσε να υπάρχει διαφορετική ερμηνεία. Το κοινό αυτό κέντρο υποστήριξης ήταν κάτι που αγωνιστήκαμε να το έχουμε στην Επιτροπή για να μπορούμε να έχουμε μια σαφέστερη αντιμετώπιση. Οι αρμοδιότητες για το ΙΤΕΡ και πέρσι με ρωτήσατε, η κυρία Γκρέσλεϊ το ζήτησε αυτό ποιος έχει την ευθύνη για ποιο πράγμα είπα ότι έδωσε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο προς τον κύριο Έτιγκερ που ήταν ένα γυαλιστερό κουτί με πλήρη ευθύνη για το ίτερ. Ο κύριος Έτιγκερ λοιπόν έχει την ευθύνη για το ίτερ αλλά θυμόσαστε ότι η αρχική πρόταση κομισιών για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές ήταν να είναι έξω από τις πολιετής προοπτικές το ΙΤΕΡ. Δεν έγινε αυτό. Αυτό είναι το οποίο είναι πολύ θετικό είναι ότι δεν βρίσκεται μέσα στον προϋπολογισμό μας. Επομένως δεν μπορεί να επιδράμει και να ληστεύει τον προϋπολογισμό της έρευνας και της καινοτομίας το ΙΤΕΡ, διότι έχει χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού, η οποία βρίσκεται βέβαια μέσα στις δημοσιονομικές προοπτικές. Αλλά ο κ. Σέτιγκερ είναι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη για το ITER. Σφάλματα. Το έθεσαν πολύ αυτό το ερώτημα. Πού βρίσκεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος σφαλμάτων και τι κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά. Αυτό το ανέφερα λιγάκι στην αρχική μου δήλωση. Έχουμε μιλήσει για το κόστος προσωπικού, έμεσο κόστος, κατανομή χρόνου. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν αναφερθεί κατ' επανάληψη από το ελεκτικό συνέδριο. Αυτή είναι η τομή διαδικασιών υψηλού κινδύνου. Γι' αυτό εμεί αγωνιστήκαμε τόσο πολύ με την υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να έχουμε την καταποκοπή απόδοση. Αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση, είχε πολλέ αντιδράσει και στο Συμβούλιο, είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά στο τέλο τη ημέρα, για να μπορέσουμε να μειώσουμε το ποσοστό σφαλμάτων, υπήρξε γενική συμφωνία για το αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφαλμάτων στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, όπως ε, ερωτήθηκε από ορισμένου ε, βουλευτές, 41% ήταν στους, ε, στο κόστος προσωπικού, 23% σε, α, σε άλλες μορφές κόστους και 31% στο έμεσο κόστος. Εκεί λοιπόν είναι οι περιοχές υψηλότερων κινδύνου. και επίσης ετέθη ένα ερώτημα από πολλούς βουλευτές αν το 2% είναι ρεαλιστικό στόχος ή όχι ως ποσοστό σφαλμάτων. Εγώ πρέπει να πω ότι είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μπορέσουμε να φτάσουμε στο 2% λιγότερο. Μπορεί να θέλουμε να αναλύσουμε και πάλι αυτό το στόχο, όπως ξέρετε, Είχαμε μια πολύ ε, τεκμηριωμένη συζήτηση για το ανεκτό επίπεδο σφαλμάτων στο παρελθόν, αλλά δεν έχουμε καταλήξει σε κάτι και εδώ η κυρία Αντρίζεν έχει δίκιο όταν μας λέει ξανακοιτάξτε το και βρείτε αν είναι πραγματικά εφικτό να υπάρχει ποσοστό σφαλμάτων 2% ή λιγότερο. Αυτό είναι και ένα θέμα που έχει αναφέρει το ελεκτικό συνέδριο και εμείς το ίδιο και εσείς το ίδιο. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν είναι ανθρωπίνο δυνατό να κατέβουμε κάτω από το 2% και ίσως η Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν σε αυτή την ανάλυση και ξέρω ότι και το Ελεκτικό Συνέδριο έχει κάνει μια συζήτηση για τα θέματα αυτά. Αυτό το οποίο εμεί πιστεύουμε ότι έχουμε πετύχει ή θα πετύχουμε στον οριζόντα 2020 είναι η απλοποίηση που πιστεύω ότι θα συμβάλλει σε χαμηλότερο ποσοστό σφαλμάτων. Η κυρία Αντρίσεν μας είπε ότι εδώ και πολλά χρόνια λέει η Κομισιόν ότι θα κάνει απλοποίηση, αλλά επειδή εγώ εργάζομαι από το 2010 συνέχεια για την απλοποίηση, θα πρέπει να σας πω ότι σε οποιοδήποτε οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό, το πιο δύσκολο είναι να απλοποιήσει κανείς τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα πραγματικά σημαντικό σύνολο μέτρων απλοποίηση που θα το αναγνωρίσει και το ελεκτικό συνέδριο και ελπίζω ότι ο ή η, η διαδοχος μου θα μπορέσει να έρθει ενώπιον του Κοινοβουλίου και να εξηγήσει πώς αυτή η απλοποίηση έχει μειώσει το ποσοστό σφαλμάτων. Για να δω. Νομίζω ότι έχω απαντήσει στα περισσότερα ερωτήματα. Αν, Αν έχω ξεχάσει, τίποτα, ε. μπορείτε να με ξαναρωτήσετε. Ε, I think there was one question... Ναι, υπήρχε μια ερώτηση ακριβώς για αυτή την καταποκοπή καταβολή. If I could have the question. Ναι, μπορείτε να μου ξανακάνετε την ερώτηση. Ο κύριος Πίπερ μπορεί να διευκρινίσει την ερώτησή του. Ναι, το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι διατεθειμένο να δεχτεί έτσι αυτές τις καταποκοπή διορθώσεις. Δεν δέχεται αυτό το επιχείρημα ότι θα μειωθεί λέει, το επίπεδο σφάλματος και το ποσοστό ε, θα ακυρωθεί με αυτό τον τρόπο καταβολής. Και μένει μάλιστα το ελεγκτικό συνέδριο. Και αυτό είναι σύγκρουση που θα βρούμε μπροστά μας ε, τα επόμενα χρόνια. Απειλεί να μας ε, συνοδεύει αυτή η διάσταση απόψεων. Και παρακαλώ, δεν ξέρω, να τα βρούνε μεταξύ τους, να συμφωνήσουν. Να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν, να συμφωνήσουν ότι ανέχονται ένα τον άλλο, να κάνουν μια κοινή δήλωση πάντως. Κύριε Επίτροπε, στη Γενική Διεύθυνση έρευνα και Κοινοτομίας δεν κάνουμε κατά αποκοπή διορθώσεις. Αυτό που κάνουμε είναι διορθώνουμε τα μεθασμένα ποσά και αυτό. And Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μόνο και του ελεγκτικού συνεδρίου για το συγκεκριμένο θέμα, τουλάχιστον συγκεκριμένη ενότητα. Για τις καταποκοπή διορθώσεις. Αυτές πάντα προκαλούν συζητήσεις. Και από ό,τι φαίνεται διέστανται και οι απόψεις ανάμεσα σε Ελεγκτικό Συνέδριο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Μπάλκο, θέλετε να μας πείτε τίποτα με δύο λόγια. Ε, για να μπορέσουμε ως Κοινοβούλιο να διαμορφώσουμε και άποψη σχετικά. Παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ. Δύο λόγια λοιπόν για αυτή την ερώτηση. Έχω την εντύπωση ότι ο συνάδελφός σας πέτυχε διάνα με το θέμα αυτό. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Μούλτερ για τις οικονομικές διορθώσεις, να σας επιστήσω την προσοχή στο κεφάλαιο 1. Στο κεφάλαιο 1 περιγράφονται αναλυτικά τι γίνεται με τις ε, ανακτήσεις των ποσών, ε, όλες αυτές τις διορθώσεις. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές εξηγήσεις. Uh, και αυτά όλα πρέπει να τα διαβάσετε πλάι-πλάι με το κείμενο της Επιτροπής και που εξηγεί πώς απαντάει. δεν περιλαμβάνονται ούτε οι διορθώσεις, ούτε το αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος. Λαμβάνονται μόνο υπόψη οι ανακτήσεις και οι διορθώσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να προσθέσει τίποτα σε αυτό και η κυρία Επίτροπος, διότι το συζητήσαμε με το προσωπικό της. Ε, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως μάλιστα. Το ελεκτικό συνέδριο καθορίζει τα κατώτατα όρια ε, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε αυτό το ποσοστό σφάλματος. Επειδή ο έλεγχος είναι συλλογικό έργο, θα ήθελα να δώσω και το λόγο στους συναδέλφους ε, οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά και κάνουν ελάχους. Ο κύριος Σούλβανης, για παράδειγμα σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε στην κυρία Γιάννη Λασέντερ και στον εισηγητή τον κύριο Πίπερ και κατόπιν θα αναλάβει τα ενία ο επικεφαλής του τμήματός μας. Ευχαριστώ πολύ. Για να πάμε στο ποσοστό των 49% των συναλλαγών με σφάλματα, τον οποίο διαπιστώσαμε για το 2011 και το 2012. Να διευκρινίσω ότι αυτό είναι το ποσοστό των συνολογών που είχαν ένα ή περισσότερα σφάλματα, τα οποία μπορεί να ήταν και ποσοτικά, μπορεί και όχι. Μπορεί να είναι ε, μεγαλύτερα ή μικρότερα ποσά τα οποία ζητούνται και εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουμε αυτά τα σφάλματα και τι ποσοστό αυτών των σφαλμάτων πηγαίνει στο ποσοστό σφάλματος. Το ποσοστό σφάλματος είναι 3,9% και αυτή είναι η καλύτερη εκτίμηση ε, σφαλμάτων τα οποία μπορούμε να σωτοκοπήσουμε και έχουν κυλικές συνέπειες. Έχουμε και ε, κάποια σφάλματα που είναι κάτω από το 0,5% η ε, συνεισφορά τους και αυτά δεν τα προσμετρούμε καθόλου. Το γεγονός ότι η συχνότητα του 2012 και του 2011 ταυτίζονται δεν θα ήθελα να πω ότι είναι τυχαίο αλλά αν δείτε τον πίνακα ε, είναι λίγο περίεργο. Έχουμε 49% τη μια χρονιά και 49% τη δεύτερη. Ε, υπήρχε όμως η, η νέα μεθοδολογία. Το 2012 λοιπόν έχουμε νέα μέθοδο που λαμβάνει υπόψη ε, κάποια στοιχεία μόνο στο σημείο της εκαθάρισης, αλλά δεν έχουμε εξήγηση για τις συνέπειες που έχουμε και γιατί έχουμε το ίδιο ποσοστό το 2011 με την παλιά μεθοδολογία και 49% και πάλι το 2012 με τη νέα μεθοδολογία. Και να πω και δύο λόγια για τις διορθώσεις. Όπως είπε και ο κύριος Μπάλκο, οι διορθώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στο ετήσιο ποσοστό σφάλματος που υπολογίζει το ελεκτικό συνέδριο. Είναι διορθώσεις οι οποίες προκύπτουν από τους εκ των υστέρων ελέγχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε λαμβάνονται υπόψη στο αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι στο υπόλοιπο ποσοστό σφάλματος. Και επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο και στον επικεφαλής του τμήματός μας, τον κύριο Γκάρντι. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχω και πολλά να προσθέσω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος. Για το 49% λοιπόν αυτή τη συχνότητα σφάλματος, που όπως σας είπαμε είναι το ποσοστό των συναλλαγών που έχουν σφάλματα. Ε, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει άμεση σχέση με την αλλαγή της μεθοδολογίας. Κατά την άποψή μου είναι η συνήθις κατάσταση αυτή. Αν λάβουμε υπόψη και την αλλαγή της μεθοδολογίας, το τοπίο όσον αφορά τις παρατυπίες δεν έχει αλλάξει από τη μια χρονιά στην άλλη. Και για να προσθέσω και σε αυτά που είπε ο κύριος Μπάλκο, για την εφαρμογή της μεθόδου που χρησιμοποιούμε, για τις διορθώσεις και τα λογιστικά πρότυπα που χρησιμοποιούμε, να σας παραπέμψω στο παράρτημα 1 του κεφαλαίου 1 της έκθεσης, το οποίο νομίζω ότι δίνει μία αναλυτική εξέγηση της μεθόδου που εφαρμόζουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτές τις διευκρινήσεις. Κυρία Επίτροπε, μπορείτε να μας παρουσιάσετε την απόψη της Επιτροπής. Μα δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ ημών και του ελεκτικού συνεδρίου για το θέμα αυτό, αλλά θέλω να απαντήσω σε ένα σημείο που ετέθη η καθυστερήσει στις πληρωμές. Είχαμε στόχους <clears throat> στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 για την προχρηματοδότηση 45 ημερών ο στόχος μας για τον ορίζοντα 2020 είναι να κατέβουμε στις 30 μέρες και για τις άλλες πληρωμές ήταν 105 μέρες και έχουμε ένα νέο στόχο στον ορίζοντα 2020 90 ημερών. Νομίζω ότι όλα αυτά πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίλντορ θέλει να πει κάτι. Τώρα καταλαβαίνω καλύτερα τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικό στα ε, δημοσιονομικά θέματα και το ελεκτικό συνέδριο ξέρει περισσότερα από μένα. Αλλά δεν βοηθάει πολύ να αλλάζει κανεί τη μεθοδολογία από το ένα χρόνο στον άλλο. Το καταλαβαίνω ότι ήταν απαραίτητο, αλλά κάνει πολύ πιο δύσκολο να συγκρίνουμε τα ποσοστά σφαλμάτων από το ένα χρόνο στον άλλο. Και δεν ξέρω, δεν έχω πάρει απάντηση στο ερώτημα του αν λαμβάνεται υπόψη η το στοιχείο των δημοσιονομικών διορθώσεων. Αν έχετε ένα ποσοστό σφαλμάτων 4% ε, και μετά ακολουθούν διορθώσεις, εγώ περιμένω να υπάρξουν ε, μικρότερα σφάλματα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δίνετε μονάχα το σφάλμα μετά τις διορθώσεις. Αλλά ίσως μπορείτε να με, να πείσετε ότι είναι καλύτερη διαδικασία που ακολουθείτε. Ακολουθεί η Ίνες Αγιάλα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, Επίτροπο για τις πληροφορίες για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό αφορά όλο το πρόγραμμα ή αναφέρατε κάποια διαδικασία για να μειώσετε την καθυστέρηση κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερη δυσκολία για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους όταν έχουν πάνω από τρεις μήνες καθυστερήσει στις πληρωμές. Αυτό είναι το ένα ερώτημά μου και το δεύτερο σε σχέση με τους ιδιαίτερους τομείς. Είπατε ναι και νομίζω ότι πολύ σωστά τα έχετε κάνει αυτά για το ίτερ αλλά βγαίνει το ίτερ το οποίο ήταν η μάστιξ του Θεού για τον ερευνητικό τομέα λόγω της πολυπλοκότητός του και του μεγέθους του και έρχεται περάσει τώρα σε ένα τομέα που τα πράγματα είναι πιο εύκολα να ελέγξετε την πολυπλοκότητα. Τώρα που έχει βγει το ίτερ από την έρευνα, Ποιο είναι το μισό που νομίζετε ότι μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ώστε να το λάβουμε υπόψη για τις ε, δικές μας έρευνες, για τη μεθοδολογία της Επιτροπής, για τις εξετάσεις εξάντε και εξπόστηκε για το ελεκτικό συνέδριο. Ποιοι τομεί λοιπόν είναι αυτοί αφού έφυγε τώρα το ίτερ και θα ξαναγυρίσει για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση και να έχουμε εποφελέστερο έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο συνάδελφος Πίπερ έχει καλυφθεί. Μέχρι και ο κύριος Πίπερ δεν έχει πια ερώτηση. Επίτροπος παρακαλώ. Ναι, ε, θα ήθελα να απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση. Βεβαίως, κάποιοι κίνδυνοι θα υπάρχουν, όπως είπα και εισαγωγικά. Δεν μπορείς να εξαλείψεις κάθε κίνδυνο. Ιδιαίτερα στις διοικητικές δαπάνες, το κόστος προσωπικού είπαμε. Έχουμε κάνει πολλά βήματα στο νέο πρόγραμμα για να προσπαθήσουμε να τα περιορίσουμε όσο γίνεται, τα σφάλματα αυτά και τα ρίσκα. Οι καθυστερήσεις των πληρωμών και οι στόχοι δεν είναι μόνο για τους μικρομεσαίους, είναι για όλους τους δικαιούχους και ενεχομένους. Ο κύριος Πάλκο. Of course I would like. Ε, ευχαριστώ. Ε, ε, για τις εξηγήσεις σας ε, και τον κύριο Μόλτερ. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα θα πρέπει να το συζητήσουμε για το συνολικό προπολογισμό και τις συνολικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 178 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το ποσό που ελέγχθηκε. Και εδώ πρόκειται μόνο για 11 δις ε, ερευνητικές δαπάνες και 6 δις για την εξωτερική βοήθεια βλέπε 16-17 βαριά βαριά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ ε, που άλλαξε η ε, μεθοδολογία και αυτή η μέθοδος δείγματοληψίας ε, συναδούν με τα λογιστικά πρότυπα. Έγιναν κάποιες διορθώσεις και οποιαδήποτε, ε, μάλλον ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι εξετάζονται με συγκρίσιμη μέθοδο και ε, τα προγράμματα που είναι στη συνδιαχείριση και εκείνα που δεν είναι σε συνδιαχείριση. Ε, χρόνο με το χρόνο υπάρχουν κάποιες διαφορές, κάποιες διακοιμάνσεις, αλλά όλα αυτά θα συμψηφιστούν και θα ε, συμπεριληφθούν. Δεν ξέρω, κάποιος συνάδελφος θέλει να κάνει ε, κάποιες συμπληρώσεις ε, για να έχουμε μια συλλογική προσέγγιση του θεσμικού οργάνου. Okay. Damit Μάλιστα. Να πούμε ότι ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που μας ήρθατε για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα που σας είχαμε υποβάλει και τα ερωτήματα. Ε, με χαρά να σας ξαναδούμε. Και... Σας ευχόμαστε και ε, ε, καλή επιτυχία για όλες αυτές τις εξαγγελίες και τα προγράμματα που έχετε υπόψη σας. Στο επανειδήν λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπάλκο και τη συνεργάτες του από το ελεκτικό συνέδριο. Ολοκληρώνεται και το σημείο 3 και πάμε αμέσως χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στο επόμενο που είναι η ετήσια έκθεση για το 2012 της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων. Α, το αναβάλαμε. Ναι, αναγκαστήκαμε να το αναβάλουμε. wir... Άρα δεν έχουμε αυτό το θέμα. Ε, και ουσιαστικά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Η επόμενη θα λάβει χώρες 16 του μήνος Δεκεμβρίου. Τι ώρα? Στις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση μέχρι την επόμενη.